Λοιπόν, ε, επιστρέφουμε στις ε, ψηφοφορίες με τις ε, τρεις προτάσεις ψηφίσματος για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους. Μιλάμε για την παράγραφο 4 του ψηφίσματος. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, τώρα, δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Votazione chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται παράγραφος 7, ε, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για το ψήφισμα με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψιώνε. Έκλεισε ψηφορία. Respinta. Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν ε, είμαστε στο ψήφισμα της Ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφορία. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. Τώρα λοιπόν έχουμε το ψήφισμα πέντε ε, πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι δύο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η, τρε, η τρία, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Σε πέντε τμήματα, όλα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Για το πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο ψήφισμα για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μισό λεπτό. Ο κύριος Λαμασούρ. Κυρία... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαπραγμάτευση για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο άρχισε πριν από λίγου μήνε, αλλά μόνο στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, που θα γίνει πρώτο γύρο τραπέζι ανάμεσα στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Το ψήφισμα που μόλι ενέκρινε το Κοινοβούλιο για την πρόταση πέντε πολιτικών ομάδων που εγκρίθηκε με πλειοψηφία πέντε έκτων είναι ένα πολύτιμο κείμενο σαφέ που υπενθυμίζει τις κόκκινες γραμμές του Κοινοβουλίου για αυτή την επικείμενη διαπραγμάτευση και την ε, εντολή που επίσημα μόλις έδωσε το Κοινοβούλιο στον πρόεδρο Σούλτς και που θα χρησιμοποιήσει όταν θα συναντηθεί ε, με τους αρχηγούς ε, κρατών και κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Έτσι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσει. Είναι ευρύτατη η πλειοψηφία και θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου. Τώρα αρχίζει η πραγματική διαπραγμάτευση. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Τώρα, ε, ψηφίζουμε για το ψήφισμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Η 15 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 12 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 5. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 3 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 2 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 10 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος, μονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα ε, Γουινέα Μπισάου. Παράγραφος 21 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 22 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 23 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 26 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο ψήφισμα για το Σουδάν και τον Νότιο Σουδάν. Η ένα παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, τελική ψηφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας Περού. Η 14. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 15 με ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 16 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η 17 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε για την 10 για το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι δύο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 21. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 6 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 23 η ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 24. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 25. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 27 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 18 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 9 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά 7 αποχές απορρίπτεται, η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε για το τελική, τελική μορφή του ψηφίσματος. Ψηφίζουμε παρακαλώ έκκληση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Σάλα Φράγκα για τον ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία του κυρίου Χαουίτ. Παρακαλώ κύριε Χαουίτ. Uh, Οι διαπραγματεύσει για αυτό το θέμα έγιναν μόλις σήμερα το πρωί και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Σαλαφρέγκα γιατί ε, καταφέραμε και με τον συνάδελφο Τσίπ και τον Τέσκι να, από τους φιλελευθέρους να καταλήξουμε σε συμφωνία, σε συνενετική λύση αποσύροντας ε, την ε, φρασιολογία των τροπολογιών των σοσιαλιστών και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από εκεί που λέμε υπό το φως της συμφωνίας του 2011 και τις προτεραιότητες. Δηλαδή χωρίζουμε διαφορετικά το κείμενο σε σχέση με αυτά που έχουμε συζητήσει ε, με την υπηρεσία σας. Ζητούμε συγγνώμη. Αποσύρω το δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας κατόπιν συνεννοήσεως με τον κύριο Σαλαφράγκα και ζητώ από τον Ολομήλα να υποστηρίξει το πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε λοιπόν κατόπιν τούτου. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το τελική ψηφορία, για το ψήφισμα, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο ψήφισμα για τις ε, διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη του ΙΕ όσον αφορά το εμπόριο όπλων. Τροπολογία 12 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 3 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίθηκε. Η 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 5 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Η 6 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 7 και η 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε οι 8 και οι 11 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 9 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα, ε, αιτιολογική σκέψη F. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα, ψήφισμα σχετικά με τις ε, εκλογές ε, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές.